τις συστάσεις των συντονιστών. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει λοιπόν από την χθεσινή μας συνεδρίαση. Χθες το βράδυ στείλαμε τα συμπεράσματα. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται δεκτές. Και θα περάσω χωρίς καθυστέρηση στις ψηφοφορίες. Είσαστε έτοιμοι. Έχουμε καταρχάς την πρόταση γνωμοδότησης του Έρνεστ Μαραγκάλ, ο οποίος δεν είναι εδώ. Α, όχι, εδώ είναι, συγγνώμη, δεν τον είχα δει, είναι στο βάθος. Για την ενίσχυση της θέσης των κοριτσιών στο σύστημα εκπαίδευσης. Αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Γυναικών. 23 Μαρτίου είχε συζητηθεί το θέμα, 30 Μαρτίου κατετέθησαν οι τροπολογίες. Δεν ξέρω, ο κύριος Μαραγκάλ θα ήθελε κάτι να μας πει πριν από την ψηφοφορία ή να ξεκινήσουμε αμέσως. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Okay. Allora, cominciamo. Partiamo allora dal compromesso 1. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Περνάμε στην τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 12 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15. Υπέρ. Κατά δεκτή. 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 18 υπέρ, κατά, δεκτή. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 τώρα. Έχει αποσυρθεί 22, συγγνώμη. 25 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25 Λοιπόν, ξεκινάμε. Πέρας ψηφοφορίες ψηφίσατε όλοι. una svista mia <laughs> approvato scusate allora eh, andiamo al 21 περνάμε στην 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά Αποχές. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβιβαστική 3. Chiusa la Τέλος. Δεκτή. Με μία ψήφο διαφορά. Περνάμε στην 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ α, κάτι δεν είπα α, μου ξέφυγε λοιπόν πάμε πίσω στην 32 κατά διέρεση ψήφος το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ δεκτή δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα 33. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 34. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 35. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 36. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 37. Κατά διέρεση ψήφος. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Για το δεύτερο τμήμα της 37. Ψηφίζεται.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 γιατί υπήρχε μια αντικατάσταση, λέει η πρόεδρος, τελικά απερίφθη. Κάποιος ψήφισε, κάποια ομάδα ψήφισε με μία ψήφο επιπλέον, ως εκ τούτου, εν πάση περιπτώσει, απερίφθη. Andiamo all'emendamento. Ecco, allora, 38. 38 διακόπτη η Πρόεδρος. Λοιπόν, ε, απερίφθη όπως είπα η προηγούμενη, γιατί η συνάδελφος που μόλις έφτασε είχε ήδη αντικατασταθεί, οπότε δεν μπορούσε να ψηφίσει και γι' αυτό και δεν ψήφισε. Θέλησε να ψηφίσει αλλά δεν είχε τη δυνατότητα. Τώρα λοιπόν, ε, οι αριθμοί των ομάδων είναι σωστοί, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, η συνάδελφος δεν ψήφισε γιατί ο αντικαταστάτης του είχε ψηφίσει. Θέλετε να γίνει μια επιπλέον ψηφοφορία αν θέλετε. «38 τροποποιημένη με την προφορική 1» υπέρ, κατά, δεκτή, 39, υπέρ, κατά, δεκτή. 40 τροποποιημένη από την προφορική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος για την πρόταση γνωμοδότηση στο σύνολό της. Υπέρ. Α, συγγνώμη, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, 22 υπέρ, Δύο κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μαραγκάλ. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη πρόταση του Ιλχάν Κιουτσούκ για την ανταγωνιστική αγορά εργασίας του 21ου αιώνα. Περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτός. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προφορική 1 Τροποποιημένοι δηλαδή 5, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 9 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 10 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμ, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 24 τροποποιημένη με την προφορική 2, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2 με προφορική. Για την 2 με προφορική. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38 Πέραστης της ψηφοφορίας. Με μία ψήφο έγινε, διαφορά έγινε δεκτή. Περνάμε τώρα στην 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψήφος με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ πέρα της ψηφοφορίας 22 υπέρ 4 κατά καμία αποχή συγχαρητήρια στον κύριο Κιουτσούκ και στο Σκιώδης. Στην παρούσα φάση λοιπόν θα περάσουμε alle, alle proposte di opinione. Allora. Στις προτάσεις γνωμοδότησης. Eh, mm, allora, cominciamo subito alle rapporti presentati da... Eh, Από τους συναδέλφους λοιπόν, τον συνάδελφο Σντροιεύσκη. για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2016 όπως γνωρίζετε. Ξεκινάμε την ε, πρόταση για την εντολή εισηγητής ο κύριος Δρογεύσκη. Η Επιτροπή θα καταθέσει την πρότασή της στο τέλος Μαΐου και η τελική ψηφοφορία λομέλια τον μήνα Ιούλιο. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Σντρογεύσκη και μετά στους κοιόδης εισηγητές. Shadow rapporteur e quindi poi i colleghi che E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα αυτό που έχω να παρουσιάσω και το εκφράζω με αδρές γραμμές, με προτάσεις τις οποίες πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι θα μπορούσατε κι εσείς να υιοθετήσετε στη συζήτηση και να συμμετάσχετε. Πέντε κύρια σημεία έχει γνωμοδότηση. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με, την, ε, με τον ήχο από τη γερμανική καμπίνα. Η γερμανική καμπίνα δουλεύει, αλλά φαίνεται ότι δεν περνάει ο ήχος. Λοιπόν, συνεχίζω. Ξεκινώ αργά-αργά για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε, αν και δεν θα σας ξεφύγει τίποτα. Πέντε κύρια σημεία λοιπόν έχει. Καταρχάς, ε, μία έκκληση. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρεκοδοτούνται με τους πόρους που χρειάζονται. Διότι το χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων υποχρεώσεων και των χρημάτων που πράγματι διατίθενται έχει σαν συνέπεια να μην υλοποιούνται καθέτος όλα τα προγράμματα. Και ιδιαίτερα θέλω να σημειώσω ότι μπορεί αυτό να πλήξει ως φαινόμενο νέα προγράμματα μεταξύ των ε, προγραμμάτων και του, και του Erasmus Plus και απευθύνω έκκληση στα θεσμικά όργανα να μην πληγεί η δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα αυτά. Προσπαθώ να επισημάνω δε στη γνωμοδότηση τα πιο ευάλωτα προγράμματα. Δεύτερον, η ανακοίνωση για την ε, ε, τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και το ρόλο τον οποίο μπορούν να δραματίσουν. Εγώ δίνω έμφαση τόσο στους τοπικούς σταθμούς όσο και στους εθνικούς εθνικής εμβέλειας. Δεύτερον, αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην πολιτιστική διπλωματία που μπορεί να αναπτύξει σε σχέση με γειτονικές χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε μια στρατηγική ώστε νέοι καλλιτέχνες, γενικά νέοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολιτιστικά προγράμματα. Επίσης, συμπληρώνω στο σημείο αυτό κάτι το οποίο έχετε ζητήσει πολλοί συνάδελφοι. Ότι δηλαδή πρέπει να προάγονται τα πολιτιστικά προγράμματα τόσο μέσα όσο και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, ε, υπογραμμίζεται η ανάγκη με προσεκτικό τρόπο να γίνεται η αναθεώρηση της χρηματοδότησης για μικρά σχέδια ή έργα ε, υποδομής ώστε οι περικοπές οι ενδεχόμενες που τα αφορούν να μην πλήξουν και τον χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι αντί να χτυπάμε κατάμουτρα στους ανθρώπους στην πόρτα να κοιτάμε προσεκτικά έχει κάποια δυνατότητα ε, να συνεχιστεί η χρηματοδότηση παρά τους ε, περιορισμούς τους δημοσιονομικούς. Και πέμπτον ζητώ μέτρα δημοσιονομικά για την καταπολέμηση της πάρα πολύ ψηλής ανεργίας των νέων, ένα πρόβλημα που επανέρχεται και είναι πάντα επίκαιρο. Επίσης παραπέμπω και στις συστάσεις ε, και τις θέσεις που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη της χρηματοδότησης του Ταμείου για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας των Νέων και του προγράμματος Juncker που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όπως σημειώνω και τα θέματα του πολιτισμού και το χώρο του πολιτισμού και τομείς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν ε, θετικές ε, διεξόδους για ανάπτυξη. Πάντως, ένα θετικό μήνυμα που μπορώ να αποστείλω είναι ότι το σχέδιο Juncker φαίνεται να λαμβάνει περισσότερον υπόψη το αίτημα και την έκκληση για τον πολιτισμό και τη συμπερίληψή του, γιατί τουλάχιστον εκεί γίνεται μια αναφορά στον πολιτισμό, ότι θα τα μεταρχικά σχέδια της Επιτροπής, και όπως είπα, θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία τον τον Ιούνιο, Ιούνιο και μετά θα πάμε στην ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ποιος ζητάει το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι. κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και νομίζω ότι θα είναι καλό για το θέμα της επικοινωνιακής ε, πολιτικής. Αναφερθούμε και στο δίκτυο Euronet, ότι δηλαδή θέλουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση του δικτύου Euronet. Είναι κάτι, βεβαίως το έχουμε ζητήσει και πάλι, αλλά θα είναι καλό η Επιτροπή Πολιτισμού να ζητήσει απερίφραστα αυτή την ε, ε, κάλυψη του δικτύου Euronet, δηλαδή να μην υπάρξει εις βάρος του κάποια εξέλιξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότησή του. Και επίσης πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την υλοποίηση του Erasmus Plus, γιατί άκουσα κάποια, ε, κάποιες αναφορές και περιπτώσεις πρόσφατα ως προς, το εκπαιδευτικό, στον, προς τον εκπαιδευτικό κλάδο του Erasmus Plus, ότι μόνο μεγάλα εκπαιδευτικά σχέδια και έργα χρηματοδοτούνται, όχι τα μικρότερα. Αυτό όμως είναι εις βάρος μας, γιατί σημαίνει ότι ε, φτάνει τελικά το πρόγραμμα μόνο σε λιγότερους ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλουμε θέλαμε λοιπόν να ανατραπούν οι ισορροπίες εκεί και θέλουμε και μικρότερα σχέδια για τα σχολεία να μπουν στην εστίαση, στην προσέγγιση και όχι μόνο τα μεγάλα. Μόργανο. che io ricevo è questo, mi scuso, non ho seguito io l'ordine. Eh, με συγχωρείτε. Εντάξει, α είναι, αφού είναι τόσο υποτικό ο κύριο Μόργαν, να ακούσουμε την κυρία Φερχάιεν. Λοιπόν, ναι. Ναι, γιατί θέλαμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στους Σκιώδης. Εφόσον συμφωνείτε κύριε Μόργαν έτσι δίνουμε το λόγο στην κυρία Φερχάιεν. Ναι, και σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά ακριβώς που είπε η κυρία Τρίπλ για την ε, διαρθρωμένη χρηματοδότηση του Erasmus ε, Plus. Το Euronet Plus, το Euronet Plus ε, δεν είχε υπαχθεί σε μια διαρθρωμένη χρηματοδότηση και νομίζω ότι τώρα πρέπει να ζητήσουμε να συνεχιστεί με έναν τρόπο σωστό και διαρθρωμένο. Η ανάγκη υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Δραγεύσκη, μικρή και μεσαίας εμβέλειας ραδιοφωνική σταθμή χρειάζονται υποστήριξη, δεν πρέπει να τους λησμονήσουμε. Στην υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο την εκπαίδευση, αλλά γενικότερα να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μία τάση να χρηματοδοτούνται τα μεγάλα, τα πιο προβεβλημένα προγράμματα και έργα και τα μικρότερα να μένουν στο περιθώριο. Όμως η διάχυση που μπορεί να έχει ως προς τον αποδέκτη και την τελική ενημέρωση αυτό το πρόγραμμα βελτιώνεται σημαντικά όταν ε, καλύπτει και τα μικρότερα προγράμματα και έργα. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να συνεχιστεί στα μικρά και μεσαία προγράμματα και όταν έρθει η ώρα για την υλοποίηση πρέπει η κατάλληλη έκθεση από πλευράς μας να, υπογράψει, να υπογραμμίσει τις διαθέσεις μας. Νομίζω ότι και στο πλαίσιο του προπολογισμού πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε χρήματα να υπάρχουν διαθέσιμα και για τα μικρά έργα και σχέδια. Ευχαριστώ τώρα ο κύριο Μόργανο. Ε, Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον εισηγητή για την εισαγωγή του και να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους που πήραν το λόγο με τους οποίους συμφωνώ. Ε, στην πρότασή του ο εισηγητής διευκρινίζει τα κομβικά σημεία για τον προϋπολογισμό του 16 και νομίζω ότι μπορούμε να τα στηρίξουμε και σε πολιτικό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να είναι συνεκτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της κατάρτισης για να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρώπης. Οι τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσω θα συμπληρώσουν το κείμενο. Σαν παράδειγμα τώρα, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο το ότι δεν θα πρέπει πλέον να ξαναβρεθούμε ξανά σε αυτήν την απαράδεκτη αναντιστοιχεία των υποχρεώσεων με τις πληρωμές για προγράμματα σημαντικά όπως το Erasmus Συν. Και επίσης μια τέτοια κατάσταση όπως είπα είναι απαράδεκτη, είναι κάτι το οποίο προκαλεί βλάβες στις οικογένειες και στα παιδιά και για την ίδια την εικόνα της Ένωσης. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ε, ευκαιρίες για να χάσουμε περαιτέρω αξιοπιστία. Ένα άλλο θέμα αφορά το ΕΦΣΙ, το πρόγραμμα επενδύσεων της Επιτροπής. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα πρέπει να βοηθήσει και προγράμματα κατάρτισης, έρευνας, ανάπτυξης των ικανοτήτων στον τομέα των ψηφιακό και στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας, ένα θέμα το οποίο η Πέτρα Κάμερβερτ είχε υπογραμμίσει και συμφωνώ απολύτως το πλαίσιο αυτό λοιπόν εγώ βλέπω ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μεγάλο βάρος και ε, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα πρέπει να διασφαλίσουμε την αηφορία τους θα έλεγα και την αυξημένη ποιότητά τους. Όπως υποστήριξε και η συνάδελφος Ζάβαλ θα ήθελα και εγώ να πω ότι τα κράτη-μέλη στον τομέα της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει ε, ε, να μειωθούν ακόμα περισσότερο στα πλαίσια των διορθώσεων του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό είναι ένα θέμα αρκετά ευαίσθητο, νομίζω ότι όμως θα πρέπει να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας σωστά. Για την σοσιαλιστική ομάδα αυτές οι επενδύσεις είναι επενδύσεις κρίσιμες, απαραίτητες για την ανάπτυξη και για τη στρατηγική, για μορφή επηρεασμού των εξελίξεων στο μέλλον. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμείς να πάρουμε τις αποφάσεις μας λαμβάνοντας υπόψη και το άειλο και το υλικό ε, ε, τρόπο αντιμετώπισης ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν εξαρτάται αν θέλετε και η ταυτότητά μας και οι οικονομικές μας δυνατότητες και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε, να είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να στηρίξουμε όλες τις μορφές που τονώνουν αυτό που θα λέγαμε ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και νομίζω ότι τελικά μετά από περαιτέρω συζητήσεις θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ο συνάδελφος Τόμ. Είχε ζητήσει το λόγο αλλά είναι απόν. Ο κύριος Μαραγάλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να επαναλάβω άλλωστε όσα έχουν ειδηποθεί. Συμφωνώ απόλυτα με τη Χέλγκα Τρούπελ. Τηλεγραφικά πέντε πράγματα. Πιστεύω θα συμφωνήσουμε από αυτόν στο πλαίσιο αυτής της νομοδότησης. Πρώτον, Συμφωνώ με αυτό που είπε ο συγητής, ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνεκτικότητα και να επαληθεύουμε ότι οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις υλοποιούνται. Και επίσης πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχεία μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων, ιδίως για το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πεδίο. Το Εράσμος, για παράδειγμα. Εκεί έχουμε συνέχεια προβλήματα. Δεύτερο θέμα, για την εκπαίδευση. Δύο πτυχές. Όλα τα προγράμματα εντός του Εράσμους και πέραν του Εράσμους όμως, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δηλαδή, και οι πτυχές της κινητικότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά και οι διάφορες περιφερειακές ανισότητες. Επίσης, πάντα σχετικά με την εκπαίδευση, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα ξεκινήσει η αναθεώρηση της δικασίας της ε, Μπολόνια και ζητείται μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν και αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης της ε, Μπολόνια. Επίσης, πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστική διπλωματία, αυτά τα δύο πρέπει να τα συσχετίσουμε. Το είπε και ο εισηγητή. Υπάρχουν πολύ κατεπήγοντα σημαντικά ζητήματα, καταστρέφονται μνημεία τη πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν όμω και κάποιε πολιτικέ προστασία πολιτιστικής και πολιτισμικής ε, κληρονομιάς και διπλωματία σε σχέση και με τρίτες χώρες των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά κινδυνεύει. Και σίγουρα εμείς θα πρέπει να έχουμε αυτή την προτεραιότητα. Τέλος, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη μεταρρύθμιση των ε, δικαιωμάτων δημιουργού, των πνευματικών δικαιωμάτων. Ίσως ένα δευτερογενές αποτέλεσμα θετικό στο μέλλον, αλλά μας ανησυχεί προς το παρόν, είναι τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αν μπορούμε να στηρίξουμε δηλαδή τους νέους ευρωπαίους παραγωγούς, ε, τις νέες καλλιτεχνικές παραγωγές. Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά. Να πω επίσης πριν κλείσω ότι θα πρέπει να προασπίσουμε, να επρασπιστούμε τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση και την πολιτισμό στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Ευχαριστώ. Ε, Βρήκα τη συνάδελφο Τόμ, αλλά την ξανάχασα. Λυπάμαι. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν υπάρχει κάποιος και από εκεί. Ε, να πω κάτι μόνο. Ε, ε, εγώ εξετίμησα το περιεχόμενο της ε, εκθέσεώς σας και να πω ε, δύο πράγματα. Να πω ότι το 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το νέο Ταμείο Εγγυήσεων για τα προγράμματα αυτά, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα για την Δημιουργική Ευρώπη Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τρέλος του 2015 θα πρέπει να δημοσιεύσει την πρώτη εκδήλωση ε, ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να προκαλέσει έτσι την προσοχή και των μεμονωμένων πολιτών και των μικρών συλλόγων και των σχολείων που ε, το θέμα αυτό τα αφορά σε σχέση με τις διδημοποιήσεις σε εισαγωγικά με άλλες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα ε, υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουν. Εμείς θέλουμε ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας ε, να υπάρξει μια κάποια ισροή πιστώσεων για να δώσουμε νέα, νέα δύναμη αν θέλετε στο θέμα της στρατηγικής επικοινωνίας. Συμφωνώ επίσης και με τη, τα θέματα της μεσαίας και μικρής κλίμακας των διαφθρωτικών ταμείων στα πλαίσια της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης του προγράμματος αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Έχω ήδη μιλήσει με τον κύριο Σδρογεύσκη σχετικά με το όριο των 5 εκατομμυρίων. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Μπορείτε να κλείσετε τη συζήτηση κύριε Ντροζιεύσκη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου για όλα τα σχόλια, σε όλους τους συναδέλφους. Υπήρξε κάτι το οποίο ακούστηκε αρκετά συχνά και είμαι ευνοϊκά διακείμενο συγκεκριμένα την ανάγκη για μια επικοινωνική πολιτική και αναφορά συγκεκριμένα στο Euronet και σε άλλα project. Αυτό είναι θετικό και το σχετίζω και με αυτό που πρότειναν οι κυρίες Τρούπελ και Κώστα. Θα περιμένω βέβαια και τις γραπτές τροπολογίες σας Είδα ότι έχει ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, αλλά να τονίσω τώρα δύο σημαντικά για εμάς θέματα. Πρώτον, ενίοτε εδώ ίσως όχι στην Επιτροπή μας τόσο, αλλά σε άλλες επιτροπές, δεν λαμβάνουμε πολύ υπόψη τα δημοσιονομικά, όπως το βραβείο Λουξ, που για μας είναι κάτι που μας γεμίζει υπερηφάνεια, όμως απειλήθηκε από μια άλλη επιτροπή και σταματώ εδώ, δεν λέω κάτι παραπάνω. Σας ε, παρακαλώ λοιπόν κυρίες και κύριοι να προσέχετε πάρα πολύ τα δημοσιονομικά ώστε και η Επιτροπή Πολιτισμού να μην χάσει το έδαφος της και τη σημασία της. Σίγουρα ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τον προπολογισμό, που μπορεί να είναι αντικείμενο βέβαια άλλων επιτροπών περισσότερο. Να πω Κατά δεύτερον, ότι διατέλεσα επί σειρά ετών Υπουργό Πολιτισμού. Και είναι απαράδεκτο, ιδίω αυτό το τόσο ευαίσθητο τομέα τη εκπαίδευση, να μην εκπληρώνονται οι δεσμεύσει και οι αναλήψει υποχρεώσεων να μην υλοποιούνται. Γιατί αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί προβλήματα. Αυτή, αυτό το κενό, αυτό το χάσμα είναι κάτι πολύ πρακτικό. Θέλω να πω επίση ότι το γεγονό ότι δεν υπάρχει εκπρόσωπο τη Κομισιόν είναι ανησυχητικό. Ελπίζω, είμαι αισιόδοξο ότι παρόλα αυτά θα ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να έχει έναν εκπρόσωπο την επόμενη φορά να μα απαντήσει. Θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχει κάτι να απαντήσει για το θέμα αυτό. Είναι ένα αίτημα το οποίο και εγώ θα ήθελα να συμμεριστώ. Συμμερίζω μάλιστα και την έκκληση του εισηγητή και του κυρίου Μόργανο για το γεγονός ότι η Επιτροπή μας πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο στα θέματα του προϋπολογισμού. Έχουμε το Europa Creative, έχουμε το Erasmus, που έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ καλά και τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν όμως κάποιες φωνές που έχουν ε, εγερθεί προκειμένου να ζητήσουν την περικοπή ακόμη και των σχετικών κονδυλίων. Πρέπει λοιπόν να, να ανακοινήσουμε το θέμα και να διεκδικήσουμε τις ε, τη διαφύλαξη στην Επιτροπή μας αυτών των αρμοδιοτήτων, το ίδιο και για το Λουξ, το, στο οποίο συμφωνούμε με τον Πρόεδρο Ταγιάννη. Και σε άλλα ζητήματα, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι απέναντι στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένε φορέ οι ομάδε δεν είναι μεταξύ του σύμφωνε. 12 Μαΐου λοιπόν στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για κατάσταση των τροπολογιών. Καλή δουλειά σε όποιον ασχοληθεί. Και περνάμε στο επόμενο θέμα με την αρφό Σουετρόβα, Σόιτροβα. Έχει την έκθεση λοιπόν. Το Μάρτιο σας θυμίζω είχαμε κάνει μια ενδιαφέρουσα ομάδα εργασίας, ένα workshop που είχαμε συζητήσει για τα θέματα αυτά τη εκπαίδευση. Τη δίνω το λόγο μετά στου και ηγητές και τους λοιπού συναδέλφου με τη σειρά. 14 Ιουλίου είναι η ψηφοφορία, κατάθεση τροπολογιών ω την 3η 12 Μαου στι 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την έκθεση που μου ανατέθηκε. Μια έκθεση που πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κατάρτιση λοιπόν, η εκπαίδευση επιχειρηματικότητα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα χρόνο ε, και μέσα στα εκπαιδευτικά συστήματα. ένας τομέας ο οποίος βοηθάει τους νέους να ξεπεράσουν προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό τους βίο, κυρίως προβλήματα σχετικά με την απασχόληση και την απασχολησιμότητα. ίσως να μην αναγνωρίζετε πάντα η σημασία της επιχειρηματικότητας και του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος, ωστόσο θα πρέπει να αναγνωριστεί ε, τόσο στα εθνικά όσο και στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι μελέτες που έχω μελετήσει δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί και να διδαχθεί. Άλλωστε αυτό μας είπε και το workshop εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να διδάσκεται, πρέπει να μαθαίνετε. Αυτό το αποδεικνύουν όχι μόνο μελέτες, αλλά και η πρακτική εμπειρία. Από διάφορα ε, ε, σχέδια μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν συνεργαστεί με σχολεία και μας καταγράφουν την εμπειρία τους. Η έκθεση λοιπόν είναι καταρμημένη σε διάφορα τμήματα στο πρώτο συνοψίζει τα έγγραφα βάσης στα οποία έχουν στηριχθεί η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, ψηφίσματα και λοιπές προτάσεις που έχουν εγκριθεί. Αυτό προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται διαρκώς ιδέες αποδεκτές. Συνοπτική λοιπόν παρουσίαση των εγγράφων και των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένη αρμοδιότητα. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να εμπλακεί και να νομοθετήσει τα θέματα ε, εκπαιδευτικά που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία σε ορισμένου τομεί και να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Σε αυτό λοιπόν μπορούμε να εντάξουμε την έννοια τη επιχειρηματικότητα στο διδακτικό πρόγραμμα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογραμμίσει τη σημασία τη εκπαίδευση, τη διδασκαλία τη επιχειρηματικότητα έτσι ώστε αυτή να προαχθεί, να μπει μέσα στο πρόγραμμα Erasmus+, έτσι ώστε να προετοιμαστεί και ένα πλαίσιο για το για προσεχές διάστημα μετά δηλαδή το 2020 γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός ε, έργων για μετά το 2020, ήδη γίνεται ο σχεδιασμός δηλαδή. Και εγώ θέλω να είμαστε έτοιμοι για την περίοδο μετά το 2020, τόσο εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε μια προοπτική για το μέλλον, προοπτική για τη δασκαλία της επιχειρηματικότητας, και αυτή είναι μια φιλοδοξία την οποία πρέπει να έχουμε. Τονίζω φυσικά ότι αυτή η διδασκαλία δεν θα κάνει κανέναν επιχειρηματία, αλλά δείχνει πώς μπορεί να αξιοποιήσει την ε, ε, δημιουργικότητά του, πώς μπορεί να αξιοποιήσει δυνατότητες ε, ανεξαρτησίας, να δώσει διάφορες ιδέες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υποστηρίζουν τα σχολεία μέσα από τα προγράμματα αυτά δεξιότητες που μπορεί να έχουν οι νέοι, να τους προετοιμάσουν για το πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο ή και για την τριτοβάθμια ε, εκπαίδευση να μπορούν να είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις επιχειρηματικότητας. Ευχαριστώ πολύ τους αδέλφους, ε, ιδιαίτερα την Κορίνα που με βοήθησε στη σύνταξη της εκθέσεως και περιμένω να ακούσω προτάσεις και συστάσεις των συναδέλφων, ελπίζοντας ότι θα είναι με τις δικές σας βελτιώσεις καλή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για την παρουσίαση. Είναι μια πολύ καλή βάση και δίνω το λόγο στον κύριο Ντράγκητσι ως πρώτο σκιώδη. Yes, uh, good morning, dear colleagues. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου με το σχέδιο έκθεσης της κ. Σοϊντρόβα. Είναι πολύ καλή δουλειά της. Όπως γνωρίζετε η επιχειρηματικότητα είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για όλους και αυτό περιλαμβάνεται και στην πολιτική στρατηγική σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω και να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτιση νεολαία για να καταστεί μια από τι σημαντικότερε δεξιότητε που πρέπει να διαθέτουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Πρέπει να ε, κατανοήσουμε ευρύτερα την έννοια αυτή τη επιχειρηματικότητα. Χαίρομαι που η συγκήτρια λέει ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε έναν ευρύ ορισμό των βασικών ε, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο τη επιχειρηματικότητα, όπω ορίζεται στο πλαίσιο του 2006 για τη διαβίου μάθηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε σε αυτή την ευρύτερη εικόνα περί επιχειρηματικότητας, γιατί είναι μια δέσμη στάσεων, συμπεριφορών, γνώσεων, δεξιοτήτων που ε, χρησιμοποιείται για διάφορους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, όχι μόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης και μπορεί να βοηθήσει ε, την ε, ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση κτλ. Βέβαια σε κάποια σημεία περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της επιχειρηματικότητας γιατί αναφέρεται μόνο σε δεξιότητες και όχι ικανότητες και γιατί δίνει έμφαση περισσότερο στο ρόλο που μπορεί να έχει ως προς την επίτευξη οικονομικών στόχων, δηλαδή άνοιγμα νέων αγορών, βελτίωση παραγωγικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η δική μας θέση είναι ότι ναι, η επιχειρηματικότητα είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξη και δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας και μπορεί να επηρεάσει θετικά ε, την προσωπική ανέλυξη και εκπλήρωση. Άρα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει πιο ευρύς ο ορισμός και το πεδίο το πεδίο και το εύρος αυτής της ε, έννοιας της επιχειρηματικότητας για να λαμβάνει υπόψη και την προσωπική και την κοινωνική διάσταση και όχι μόνο την οικονομική. Γιατί έτσι Διευρύνδεται το πεδίο της επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνει τους πάντες και και αυτό θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που πρέπει να εισαχθεί στην εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε και να επικυρώσουμε τις ικανότητες και την άτυπη μάθηση μεταξύ αυτών καταπολέμηση ανισοτήτων στην εκπαίδευση, ιδίω για του νέου που ανήκουν σε μειονεκτικέ ή ευάλωτε ομάδε, ε, που λόγω αυτή τη κατάσταση παρεμποδίζεται γενικώ η ανέλυξή του και η ευημερία του. Πρέπει να έχουμε επίση εταιρικέ σχέσει, διατομιακή συνεργασία και ένα συνεπέ εθνικό ε, και ευνοσιακό πλαίσιο πολιτικό και μέτρων. Με την κυρία Σοντρόβα θα έχω συνεργασία, αλλά και με τους άλλους συζητητές για τη σημαντική αυτή έκθεση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και αγαπητοί συναλφοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Σόιντροβα για την ε, εκτεταμένη κάλυψη του θέματος. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάποιες ε, παρατηρήσεις, κυρία Σόιντροβα. το δυναμικό που έχει για προαγωγή ε, η Ευρώπη της διδασκαλίας στην επιχειρηματική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ωστόσο και εμείς να προσθέσουμε την ιδιαίτερη συμβολή της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα των νέων γιατί βλέπω σαν να έχει περιοριστεί μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης ε, η στόχευση της έκθεσης. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να στραφούμε και προς τους νέους και να ενθαρρύνουμε, να δώσουμε κίνητρα, να εμπνεύσουμε για την επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι διδάσκοντες, υπογρεμίζοντας το δυναμικό που προσφέρουν διάφορα ψηφιακά εργαλεία, δυναμικό ανάπτυξης, δυναμικό διεύρυνση των γνώσεων των νέων και της επιχειρηματικότητάς τους. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες να ξεπεράσουν τα χάσματα και τα κενά στην κατάρτισή τους. Μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε μέσα από αυτό κατάρτιση, ε, coaching, την ε, λεγόμενη υποστήριξη, φροντιστηριακή υποστήριξη και άλλες λύσεις που μπορούν να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα ένα σημαντικό δηλαδή παράγοντα παραγωγικότητας, ανάπτυξης, δημιουργίας της Η Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω δε την ανάγκη βελτίωση τη συνεργασίας και τη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πρακτικών μεταξύ των ε, κρατών μελών που έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα σπουδών τους την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας και την ανάγκη να ενθαρρυνθούν όσα κράτη δεν το έχουν ακόμη πράξει να προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ το πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από χώρες οι οποίες είναι επιτυχείς στον τομέα της επιχειρηματικότητας, βλέπουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και με θετικό τρόπο την αποτυχία, έτσι ώστε να έχει κανείς μια δεύτερη και τρίτη ευκαιρία και να μην καταδικάζεται με την πρώτη αποτυχία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. να δείξουμε ακριβώς ότι μια μορφή τέτοια αποτυχίας μπορεί να είναι και ε, δεκτή. Η Πέτρα έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για τις προτάσεις της. Σε ένα-δύο σημεία θα ήθελα να επιμείνω, ε, γιατί έχουμε παραδείγματι και στο Erasmus Plus, ένα κομμάτι που ονομάζεται Erasmus Plus Entrepreneurship, επιχειρηματικότητα. Ένα κομμάτι του προγράμματος Erasmus Plus που δεν είναι γνωστό αρκετά. Και μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ήταν καλό να διαδοθεί περισσότερο η ενημέρωση για το πρόγραμμα αυτό για να εξαντληθούν καλύτερα, να αξιοποιούνται καλύτερα οι δυνατότητες που προσφέρει. Μέρος του Erasmus πλάσου, όπως είπα, ωστόσο, αφού δεν είναι ακόμη αρκετά ε, γνωστό και όσο μας καλεί και η Επιτροπή να το προβάλλουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πτυχή αυτή, ότι υπάρχουν δυνατότητες, ότι υφίστανται δυνατότητες για αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας. Επίσης, από την ε, πατρίδα μου, μπορώ να σας ενημερώσω πως υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα από σχολικές ε, εμπειρίες, πειράματα καλύτερα, που ε, βλέπουμε σε ένα σχολείο να ξεκινάνε μια μικρή επιχείρηση. Ένα περίπτερο φερρυπίν, έναν τρόπο τα παιδιά να μάθουν στην πράξη και μαζί την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη ώστε να αναζητήσει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των νέων όπου υπάρχουν τέτοια καλά παραδείγματα. Βεβαίως θα ήθελα επίσης να επισημάνω ένα κάπως επικριτικό πνεύμα στα όσα κάνουμε, να μην λησμονήσουμε τις ισορροπίες της ε, εκπαίδευσης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να γύρει πλάστικα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στην ε, οικονομική διάσταση και θεώρηση της ε, εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε αναζητώντας έναν τρόπο να υποστηρίξουμε την οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα των εκπαιδευομένων, των μαθητών και άλλες δεξιότητες που πρέπει να προσφέρει το σχολείο όπως ε, την, ε, τις κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία, την κοινωνική και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι ακόμη, ε, δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι για να μπορέσει ένα δάσκαλο να διδάξει την επιχειρηματικότητα θα πρέπει ο ίδιο να έχει κάποια εμπειρία ή ικανότητα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Βλέπουμε ωστόσο ότι η κλασική σταδιοδρομία ενό ε, δασκάλου είναι ότι έχει περάσει από τα σχολικά θρανία, περνάει μετά στα έδρανα του Πανεπιστημίου και επιστρέφει στο, στη σχολική αίθουσα ω δάσκαλο χωρί ποτέ να έχει εκτεθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στο γεγονό ότι χρειάζεται να δούμε δούμε την πρόκληση που αντιμετωπίσει ο δάσκαλος όταν κληθεί να διδάξει την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη που θα πρέπει να του προσφέρουμε ώστε να τα καταφέρει. Πρέπει και στον τομέα αυτό να εργαστούμε. Και το θέμα είναι όχι μόνο να μπορέσουμε να προβάλλουμε την ε, οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα σαν δεξιότητα, αλλά ταυτόχρονα να εξηγήσουμε στο μαθητή, να του δώσουμε μία πρώτη γεύση για το τι σημαίνει επαγγελματικό βίο. Γιατί μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο κανεί δεν έχει καμία σχεδόν ή πολύ περιορισμένε ιδέε για το τι μπορεί να σημαίνει η ζωή στην ε, ε, επαγγελματική δραστηριότητα. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο να μπορεί κανείς να μεταβαίνει σε, μια επιχείρηση, σε μια πραγματική δουλειά εντός εισαγωγικών, ώστε να ε, βλέπει στην πράξη τι σημαίνει και έτσι να μπορεί ο δάσκαλος δηλαδή να μεταδίδει ε, τη γνώση αυτή και την εμπειρία αυτή στους μαθητές του. Ευχαριστώ πολύ Λιμπάτσικα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την κυρία Σόιντρόβα. Όχι μόνο για την εκπόνηση της εξαιρετικής αυτής έκθεσης, αλλά και γιατί ασχολήθηκε με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οκτώ μόνο ευρωπαϊκές χώρες έχουν την επιχειρηματικότητα ως εκπαιδευτική ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει και πραγματικά είμαι υπερήφανη γιατί διατέλεσα το 2002 υπουργό Πολιτισμού και εισήγαγα στην εκπαίδευση την ενότητα της επιχειρηματικότητας, το μάθημα της επιχειρηματικότητας. Δύο πράγματα είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερε και η Πέτρα, οι διδάσκοντες, γιατί ένας δάσκαλος, ένας καθητής που δεν έχει κίνητρο ε, και δεν τον ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί και να τη διδάξει. Μια από τις βασικές δραστηριότητες λοιπόν θα πρέπει να είναι η ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών μεταξύ των διδασκόντων. Θα μπορούσαμε ίσως να ε, προωθήσουμε και ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ε, ή κινητικότητα ε, των διδασκόντων στο πλαίσιο του Εράσμου σε άλλων προγραμμάτων. Και το δεύτερο είναι ένα θέμα που εν μέρει ήδη αναφέρθηκε, δηλαδή επιχειρηματικότητα, ε, είναι κάτι που πρέπει να το προσεγγίσουμε ολιστικά, γιατί δεν είναι μόνο η ίδρυση μιας επιχείρησης, είναι μια δέσμη δεξιοτήτων επιχειρηματικών αλλά και διαπροσωπικών. Δημιουργικότητα, ε, σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάλυση κινδύνων. Πρόκειται για μια ολόκληρη δέσμη δεξιοτήτων και ικανοτήτων αν δούμε έτσι την επιχειρηματικότητα, ε, τη βλέπουμε υπό τελείως διαφορετική οπτική γωνία, γιατί υπάρχουν και διάφορα στάδια της εκπαίδευσης όπου μπορούμε να τονίσουμε την επιχειρηματικότητα και από διαφορετικές πτυχές σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επίπεδο. Καταθέσουμε τροπολογίες για να τονίσουμε και τη σημασία της επιχειρηματικότητας και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, ανθρωπιστικές επιστήμες, πανεπιστήμια. Και επειδή έχω το λόγο, θα ήθελα να παρεκκλίνω λίγο από την έκθεση αυτή και να μιλήσω για κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ ευχάριστο που έχω να σας πω. Είχαμε ήδη μία πρώτη επιτυχία ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια. Μου είπαν οι υπουργοί της Μπένελουξ ότι στις 9 ε, Μαΐου θα υπογράψουν συμφωνία για την αυτόματη αναγνώριση των ε, ακαδημικών προσόντων, που ήταν ένας βασικούς μας στόχους. Να λοιπόν μια πρώτη επιτυχία. Δεν προχωρήσαμε περισσότερο στο αλλά τουλάχιστον τρεις αυτές χώρες θα προχωρήσουν σε αναγνώριση αυτών των προσόντων. Συγχαρητήρια και γι' αυτό και πάνω απ' όλα γιατί είμαι βεβαία ότι η δική μας υποστήριξη και η μεγάλη πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε το έγγραφο ήταν αυτό το, το οποίο βάρινε στην απόφαση το Αντέλη. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Την εισηγήτρια νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση. Όλοι φαίνεται εδώ ότι συνενούμε για τον ρόλο της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ πάντα αυτό προσπαθούσα να κάνω, να είμαι σωστός επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάζει κανείς τις ιδέες σε εφαρμογή. Και το θέμα δεν είναι να διαπιστώνει τα κενά της αγοράς μόνο, αλλά και τα κενά της κοινωνίας και γι' αυτό οι συζητήσεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με την κοινωνική ατζέντα ήταν πολύ χρήσιμες. Να πω ότι τα παιδιά γεννιούνται με μια φυσική περιέργεια, μια περιέργεια η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν επιχειρηματικότητα. Αν δείτε τα παιδιά να παίζουν, ε, χρησιμοποιούν συμπεριφορές επιχειρηματικότητας their interactions with other people. And I would just like us not to forget that I think this is something that can be done at a really, really early age. Νομίζω λοιπόν ότι από πολύ μικρή ηλικία μπορούμε να εμφυσίσουμε αυτή την οτροπία στα παιδιά. Πριν λίγο καιρό είχα πάει σε ένα σχολείο σε μια γεωργική περιοχή στην εκλογική μου περιφέρεια και ένας ε, παραγωγός ε, ε, κακάο από τον Μπελίζε επισκεφτόταν τα παιδιά και έφτιαχναν σοκολάτα και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αν η επιχειρηματικότητα είναι και ευχάριστη τότε θα το κάνει κανείς με πολύ μεγάλη χαρά και προθυμία. Και μαθαίνεις πράγματα, το ποιος το φτιάχνει, ποιος το πουλάει, ποιος το αγοράζει, γιατί ο κόσμος το θέλει Αυτά ε, μπορεί να τα κατανοήσει ένα νέο παιδί στα πλαίσια ακριβώς της ε, έννοιας της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Μπορούμε να βάλουμε επίσης στο μυαλό των ανθρώπων και την χρησιμότητα ε, των κοινωνικών μορφών εμπορικής δραστηριότητας όπως τα κοινωνικά ταμιευτήρια, όπως τα, οι συνεταιρισμοί οι κοινωνικές συμπαραγωγές, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία, ε, όπως και οι εναλλακτικέ εμπορικές δραστηριότητες, ε, έχουν ε, υποστηριχθεί αυτές οι δραστηριότητες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα θέλουμε τη δικαιοσύνη στο εμπόριο, πάντα θέλουμε τη δικαιοσύνη στην επιχειρηματικότητα. Είναι στόχος του Κοινοβουλίου. Απαιτείται λοιπόν να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει με τη φτώχεια στον αναπτυσσό και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις βέλτιστες δυνατές πρακτικές όπου αυτό είναι εφικτό. Σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση Νεκόβα. Ε, ευχαριστώ συνάδελφε. Οι προηγούμενοι ε, ε, που μίλησαν για την επιχειρηματικότητα είπαν πράγματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε την επιχειρηματικότητα σαν ένα ε, θα έλεγα θέμα, αλλά απλά ενδιαφέρον. Είναι κάτι το οποίο αφορά και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία και την πρωτοβάθμια ακόμα εκπαίδευση είναι πράγματα και γνώσεις που είναι χρήσιμα για την προσωπική ζωή. Δεν θα πρέπει να το βλέπουμε όμως αποκλειστικά με την οικονομική του πλευρά. Να δούμε ακριβώς τι δυνατότητες δίδει η επιχειρηματικότητα στους νέους, να δούμε ε, πώς μπορεί ακριβώς να βελτιώσει τη ζωή των εμπλεκομένων. στην Ευρώπη οι νέοι που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες αντιστοιχούν στο 37% του πληθυσμού, ενώ στο στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι το 50%. Ε, γνωρίζουμε βέβαια ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, είναι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν θέλουμε περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τέτοια θέματα, θα πρέπει να αναπτύξουμε ακριβώς την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Από την άλλη, σε οικονομικό επίπεδο πια, όταν μια χώρα ή μια κοινότητα επενδύει στην επιχειρηματικότητα, η απόσβεση είναι περίπου 1 προς 40. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πόρο οικονομικό, ο οποίος ε, θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας, ιδιαίτερα μέσω των νέων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και οι νέοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν βλέποντάς το στην πρώτη φάση σαν παιχνίδι. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε κάτι εδώ να πει, μια κάποια παρατήρηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα αυτή την πρωτοβουλία για πρόθεση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να τονίσουμε την ανάγκη αυτής της ολιστικής διακλαδικής διατομιακής προσέγγισης τη επιχειρηματική εκπαίδευση και την εστίαση στη νεολαία. Θέλουμε επίσης ε, να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι πράγματι θα πρέπει να συμπίξουμε έναν ε, ε, συνασπισμό, μια συμμαχία μεταξύ διαφόρων εταίρων και από την τυπική και από την άτυπη εκπαίδευση και μάθηση. Θα ήθελα να σας πω ότι και η άτυπη μάθηση βοηθά γιατί εφοδιάζει τους νέους με εγκάρσιες δεξιότητες και επιχειρηματικές δεξιότητες μεταξύ άλλων. Κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα αποτελεί μια πλατφόρμα ιδιαίτερα κατάλληλη γιατί μπορεί να φέρει σε δύο τραπέζι τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς για ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών, και έχουμε δει και από διάφορες εκθέσεις σε σχέση με την νεολαία ότι υπάρχουν ήδη πολλές πρωτοβουλίες για την επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά πρέπει σίγουρα να διδαχθούμε ένας από τον άλλο και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus εστιάζει ακόμη περισσότερο πλέον στην επιχειρηματική εκπαίδευση, όχι μόνο στην υπαριθμόν 1 βασική δράση, αλλά και στην υπαριθμόν 2 βασική δράση. Δηλαδή στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, διακρατικές ε, πρωτοβουλίες νεολαίας, ε, συμμαχίες γνώσης και τομεακών δεξιοτήτων και εκπαίδευση των εκπαιδευτών είναι και ένα θέμα που μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Τώρα όμως, αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου, που ίσως έχει να συμπληρώσει. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Από την πλάτη της εκπαίδευσης. Να πω ότι πράγματι υπάρχει αυτή η προσέγγιση και πρέπει να την έχουμε υπόψη και επίσης σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, δηλαδή στα σχολεία θα πρέπει να εστιάσουμε, να κάνουμε πιο επιχειρηματικά, αν θέλετε, τα παιδιά, αλλά και στον τομέα τη επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη και στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Όπω είπε η συνάδελφο, επιχειρηματικότητα ήδη ε, κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο σιάλκο. Το 2006 είχαμε και την ανακοίνωση για τι βασικέ δεξιότητε και στο Erasmus Plus ε, η επιχειρηματικότητα αναφέρεται παντού. Και νομίζω ότι και σε πολλά κράτη-μέλη είναι ένα θέμα που απασχολεί. Θα πρέπει απλά να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Μα ικανοποιεί που και σε εσά αποτελεί προτεραιότητα το θέμα τη επιχειρηματικότητα. άρα μπορούμε να σημειώσουμε προ. Έχω κάποια συγκεκριμένα σχόλια. ίσονο σημασία, οπότε θα μπορούσα να τα συζητήσω διμερώ με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Όντω ε, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ενεργό συμμετοχή στην Επιτροπή. Ξαναδίνω το λόγο στη συνάδελφο Σόεντροβα. Και τι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια. Και να σημειώσω ότι μπορούμε να τα ενσωματώσουμε σε μεγάλο βαθμό στις τροπολογίες. Προσπαθώ να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία της ε, επιχειρηματικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης σαν σύνολο, αλλά μπορούμε να κάνουμε τις ευκρινήσεις που ζητάτε. Και βέβαια τις ευκρινήσεις που αφορούν την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης μπορούμε να υπογραμμίσουμε το ρόλο του προγράμματος Erasmus Plus, που ήδη καλύπτεται στο σημείο 4, κάπως περισσότερο. Και για τις βέλτιστες πρακτικές επίσης προτείνω ένα δίκτυο που θα μπορούσε να οργανώσει η ίδια η Επιτροπή, ένα δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, κάτι τέτοιο, που θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σημειώνω λοιπόν όσα μα είπατε. σα ευχαριστώ για τα σχόλια. Θέλω απλώ να υπογραμμίσω ότι στα συμπεράσματα λέω όπως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος τη θητεία να καταθέσει μια ενδιάμεση έκθεση για τα θέματα τα οποία έχω προτείνει. Ξέρετε, είμαι από αυτού του ανθρώπου που όταν κάνουν κάτι θέλουν να βλέπουν ε, απτά αποτελέσματα. Ελπίζω λοιπόν στο τέλο τη θητεία να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ανάλυση τη αποτελεσματικότητα των προτάσεων, τη υλοποίηση του δικτύου, τη ε, βελτίωση των βέλτιστων πρακτικών ε, χάρη στο Erasmus Plus και έτσι να σε θέση πέντε χρόνια να ξαναδούμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ όλου του συναδέλφου για τη συμμετοχή στη συζήτηση και υπενθυμίζω ότι. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει την έκθεση στις 14 Ιουλίου, στη τελευταία της συνεδρίας πριν από τις διακοπές. Τροπολογίες έως τις 12 Μαΐου. 12 η ώρα το μεσημέρι και θέλω ιδιαίτερος να σημειώσω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση πάνω στην οποία στηρίζεται η έκθεση και οι επιλογές της. και από πλευρά του Κοινοβουλίου, καθώ είμαστε σε μια πρωτο, πρώτη φάση τη υλοποίηση των πολιετών προγραμμάτων. Όπω είπατε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε και για την περίπτωση του Erasmus, αλλά και για την ε, διαβίου μάθηση, το long life learning, ε, μια ανάλυση, μια μελέτη για την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας και βέβαια τον αντίκτυπο προς την απασχολησιμότητα. Ελπίζω να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και οι φυστάμενες πλατφόρμες αλλά και ε, άλλες λύσεις συνεργασίας με την Επιτροπή μας. Και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ενημερώνει πάντοτε. Μιλήσατε για μια έρευνα για 23 κράτη που έχει γίνει για το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε όμως να υπάρξει η επικαιροποίησή της και η αξιοποίηση των ευρημάτων της και ενδεχομένως ανάπτυξη δικτύων ε, σχολείων ή ανώτερων ανώτατων ιδρυμάτων στον χώρο αυτό. Είτε μέσα από το Erasmus, Entrepreneurship, Erasmus Plus Entrepreneurship, είτε μέσα από ε, άλλα έργα, μακράς πνοής θα έλεγα, ή μέσω κάποιων ε, θυλάκων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν γύρω από σχολεία ε, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και έτσι θα μπορούσαν να δώσουν τον πολλαπλασιαστικό, ε, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα τέτοιου είδους μικρά προγράμματα με τη μορφή των clusters. Ευχαριστώ. Διακόνω τώρα είναι η επόμενη έκθεση. Θέλω μόνο να σας ενημερώσω πριν ενδεχομένως αποχωρήσουν κάποιοι συνάδελφοι, αν και ελπίζω να μην αποχωρήσουν. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι αύριο και έχω ήδη ενημερώσει τον ιστές, θα το επαναλαμβάνω όμως. Αύριο, αν είσαστε εδώ παρόντες, γίνεται μια κοινή ακρόαση με πρωτοβουλία της Επιτροπής των Πολιτικών Δικαιωμάτων και κοινή με τη δική μας Επιτροπή. Αύριο, 9.30 με 11.30, στον τρίτο όροφο στην ίδια αυτή αίθουσα ε, για, τον, για το θέμα των, ε, του αθλητισμού. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Μπακού για τον αθλητισμό. Αρμοδιότητες έχουμε και εμείς στο, για τον αθλητισμό, για την προαγωγή του. Και έτσι θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με το αυριανό σεμινάριο, αλλά και να συνεχίσουμε με πολιτικές πρωτοβουλίες στο χώρο του αθλητισμού που θα θέλαμε να ενισχύσουμε. Σας ενημερώνω, θα είναι παρόν και η Πρόεδρος Βαλενσιάνου από την Επιτροπή των Δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο. Grazie. Stimați colegi, eh, comisia η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για μια γνωμοδότηση για τη συγκεκριμένη έκθεση. Η υπεύθυνη επί της ουσίας Επιτροπή είναι η Τζούρη, η Νομική Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε το θέμα ε, της, ε, των ε, σημάνσεων γεωγραφικής προέλευσης και σε άλλα προϊόντα πέραν των γεωργικών. Η συμπερίληψη τέτοιων προϊόντων θα βοηθήσει γενικά νομίζω την ανάκαμψη του βιοτεχνικού τομέα. Έχουμε πάρει κάποιες πρώτες απαντήσεις, είχαμε κάποιες πρώτες συζητήσεις, είχαμε μια συνάντηση των εισηγητών με συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εφικτό αυτής της δράσης. Βέβαια από πλευράς ε, του πολιτιστικού τομέα μια τέτοια πρωτοβουλία είναι πολύ θετική. Αλλά παρόλα αυτά απαιτείται να υπάρξει ένας καλύτερος καθορισμός του νομικού πλαισίου. Όταν μιλάμε για παραδοσιακά ε, βιοτεχνικά επαγγέλματα, βιοτεχνικές δραστηριότητες, κάτι τέτοιο θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Απαιτείται λοιπόν εμείς ε, να διατηρήσουμε στο επόμενο νομικό πλαίσιο, στο επερχόμενο νομικό πλαίσιο και το θέμα ε, της προέλευσης. Αυτό συνδέεται βέβαια και με ένα άλλο θέμα που είναι η τεχνολογική καινοτομία. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι αντιφατικό αυτό το να προστατεύσει κανείς ένα παραδοσιακό προϊόν μέσα από τις τεχνολογικές καινοτομίες. Όχι. Νομίζω ότι ε, υπάρχει μια κάποια ελευθερία σε σχέση ε, με τις βιοτεχνικές δραστηριότητες. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές αρκεί να μην θυγεί η ταυτότητα και ε, το αυθεντικό του προϊόντος. Να υπογραμμίσω λοιπόν εδώ ότι το σύστημα αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για κάποιες ε, βιοτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες επιβιώνουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Να σας θυμίσω επίσης ότι οι βιοτέχνες έχουν ανάγκη από προστασία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα εδώ, αστείο λίγο, σας το δίνω. Κοιτάξτε τι ωραία είναι αυτή η τσάντα, πώς μπορείτε να συνδυάσετε τον προηγούμενο αιώνα με τον δικό μας αιώνα. Dacă vă place Κοιτάξτε, αν σας αρέσει αυτή η ψάφινη τσαντούλα, εγώ θα πάρω ένα τηλέφωνο σε κάποιον στη χώρα μου και θα φέρω τέτοιες τσάντες για όσα λάπτοπ εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα παράδειγμα είναι μια γυναίκα η οποία το φτιάχνει αυτό στο δέλτα του Δούναβη και έχει φτιαχτεί από... η ε, ουνίτε Delta Δέλτα Și în final, iată cum se întâlnesc cele două. Aș putea, aș vrea să vă spun multe, multe lucruri. Mi se pare că este o Είναι φτιαγμένο λοιπόν από τα εξωτερικά φύλλα της, ε, του φυτού της κάναβης. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες, υπάρχουν τέτοιου είδους βιοτεχνικές δραστηριότητες και έχουμε επίσης ε, και την δυνατότητα να φέρουμε ξανά στην επικαιρότητα κάποια προϊόντα τα οποία στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και αυτό νομίζω ότι θα μας ε, ε, <clears throat> εξασφαλίσει τη συνέχεια στην ταυτότητά μας οι γνώσεις δεν θα χαθούν σε τομείς ποικίλου όπως ακριβώς και η κεραμική, ε, όπως η αλλουργία, έχουμε συγκεκριμένες ε, ικανότητες, άνθρωποι που φτιάχνουν βιτρό ε, θα χαθούν αυτές οι ικανότητες σιγά σιγά αν δεν πάρουμε μέτρα, αν δεν παρέμβουμε έτσι ώστε να μείνουν ζωντανά αυτά τα επαγγέλματα και αυτό σημαίνει και χρήμα, αυτό σημαίνει και θέσεις απασχόλησης, αλλά βασικά σημαίνει ηθική υποχρέωση από πλευράς Σας ευχαριστώ λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σας και το παράδειγμα που δώσατε. Είναι σημαντικό το θέμα. Έχει υπάρξει ένα green paper όπως ξέρετε, το οποίο εξέτασε τον τρόπο ε, με τον οποίο μπορεί κανείς ε, να προστατεύσει όπως προστατεύουμε τα γεωργικά προϊόντα και τα βιοτεχνικά προϊόντα και τα προϊόντα του πολιτισμού. Ο συνάδελφος Νεκόφ έχει ζητήσει το λόγο και άλλοι δύο συνάδελφοι μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντιακόν για την πολύ υποδομητική δουλειά του. Κατ' εμέ είναι πολύ ισορροπημένη η γνωμοδότηση, εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να διατηρηθούν ε, και τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε σχέση και με μη γεωργικά προϊόντα. Θα μπορούσε και η πολιτιστική κληρονομιά να υποστίζει με αν δεν προστατεύσουμε αυτά τα προϊόντα. Γι' αυτό και είμαι υπέρ ενός ενοποιημένου συστήματος για τις γεωγραφικές ενδείξεις μη γεωργικών προϊόντων. Αυτό θα ενθαρρύνει την οικονομική, τεχνολογική ανάπτυξη ορισμένων περιφερειών, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της παραγωγής παραδοσιακών αγαθών. Ο ε, εστίασα στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με μη γεωργικά προϊόντα και την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων. Πολλά από αυτά τα γεωργικά προϊόντα βασίζονται σε κάποιες παραδοσιακές δεξιότητες. Μιλάμε για μια πλούσια, πλουσιότατη πολιτιστική κληρονομιά, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε και να, να τα σε επόμενες γενναίες ότι αυτό αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι θα γίνουν ευρύτερα γνωστές αυτές οι δεξιότητες. Θα αναγνωριστεί δε και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αυτών των μη γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τα περιφερειακά προϊόντα για να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και για να εξασφαλίσουμε δίκαιη αμοιβή στους τοπικούς παραγωγούς. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, κατάρτιση αυτών των παραγωγών μη γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να καταστήσουμε πιο ελκυστικά αυτά τα επαγγελματα, αυτές τις τέχνες. Κατά κλείδι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν σχετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη αυτών των παραδοσιακών και επαγγελμάτων. Πρέπει να προωθηθεί επίσης ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός. Και θα πρέπει ίσως ε, να μπει και ένα μάθημα στα σχολεία. Δηλαδή στη διδακτέα ύλη να περιλαμβάνεται αυτό το αντικείμενο. Έτσι, οι σχετικέ γνώσει θα μεταφέρονται όχι μόνο σε επαγγελματίε, αλλά από γενιά σε γενιά σε όλου του πολίτε. Τέλο, Θα πρέπει αυτή η προστασία να επεκταθεί και σε, διάφορα παραδοσία, σε διάφορες παραδοσιακές διαδρομές. Στην Ισπανία που είχα πάει, μίλησα για αυτό το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων σε διάφορες παραδοσιακές διαδρομές, παραδοσιακές χάρη κεραμικά. Υπάρχουν περιφέρειες που παράγουν κεραμικά. Θα μπορούσαν να να καταστούν πιο ελκυστικέ. να αυξηθεί ο τουρισμός. Ευχαριστώ. E ευχαριστώ, Μακλόρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εμείς στο ECR ακόμη δεν έχουμε πιστεί για το πόσο χρειάζεται ένα τέτοιο μέτρο και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση για τις συνέπειες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το κόστος και τα μειονεκτήματα γιατί υπάρχει κίνδυνος αντί να ενθαρρύνουμε να ε, παρακολύσουμε την καινοτομία. Δηλαδή να πιέσουμε τους ανθρώπους προς παραδοσιακά επαγγέλματα ή τέχνες που ε, σημαίνουν ταυτόχρονα ότι θα προχωρήσουν σε κάτι καινούριο. Θέλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε μία λύση η οποία δεν θα ακολουθεί απαραίτητα τις γεωγραφικές ε, ονομασίες. Ε, μπορούμε να βρούμε λύσεις με διαφορετικά μοντέλα σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικά μοντέλα. Βεβαίως οι μη γεωγραφικές, οι ε, ονομασίες που δεν είναι γεω, γεωργικού τύπου, δεν είναι αγροτικής προέλευσης, έχουν τη σημασία τους, αλλά στο να δώσουν ε, σε ένα προϊόν αξία όταν θεωρούνταν ότι δεν ήταν ε, επαρκή η αναγνώρισή του, η αναγνωρισιμότητά του. Εμεί θέλουμε και να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων βεβαίω, αλλά και να εξασφαλίσουμε την ευελιξία ω προ τον τρόπο παραγωγή. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπου έχουν προσδιοριστεί ζώνες ακτίνας 2 χιλιόμετρων, ας πούμε, 2,5 χιλιόμετρων, πάρα πολύ μικρές δηλαδή. Ε, πρέπει να αφήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Και θα ήθελα να ξέρω πόσες από τις χώρες μέλη, εάν υπάρχουν στατιστικές, έχουν υιοθετήσει μη γεωργικής ε, πρόλευσης ονομασίες ε, γεωγραφικές. Εάν αυτό έχει κάποια σημασία φυσικά θα το διαγνώσουμε και επίσης θέλουμε να δούμε τι, τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν χρειάζεται να γίνει κάτι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να λέμε ότι α, θα προστατεύσουμε το τάδε επάγγελμα την τέχνη και θα διορθωθούν όλα τα προβλήματα. Χωρίς να χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε, υπάρχουν κάποια προϊόντα πολύ ενδιαφέροντα, όπως αυτή η θήκη για φορητό υπολογιστή που έφερε ο συνάδελφος, αλλά και στη δική μου την περιφέρεια έχουμε ωραία προϊόντα που μπορούμε να προβάλλουμε, χωρίς όμως να γινόμαστε προστατευτικοί τόσο ώστε τελικά να μην προάγονται τα προϊόντα μας. Να έχουμε το αντίθετο δηλαδή αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη σας. ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα πολιτισμικά αυτά προϊόντα που θεωρούνται για λόγους ιστορικούς για ένα έθνο σημαντικά πρέπει να προστατεύονται. Η Ουγγρική κυβέρνηση με, αυτή την, ε, με αυτό το πνεύμα προχώρησε σε μια καταγραφή ε, ουγγρικών προϊόντων μέσα σε ένα κατάλογο που έλεγε ότι αυτά είναι τα παραδοσιακά μας προϊόντα, τα προστατευόμενα. Αυτό αφορά ορισμένα είδη ε, κλώστο υφαντουργίας, ορισμένα υφαντά, κεραμικά από συγκεκριμένες περιοχές και άλλα προϊόντα. Σε ένα κατάλογο λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό από τη γεωγραφική ένδειξη. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα προϊόντα αυτά, και πιστεύω ότι πρέπει να τα προστατέψουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει προστατευτισμό. Είναι πολιτιστικά προϊόντα και πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική ένδειξη. Κυρία Τρίπελ, ευχαριστώ τον κύριο Γιακονό για την ομιλία. Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την ανάγκη να γίνει μια μελέτη σοβαρή, να καταγράψουμε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της προβολής αυτών των αυτής της διάστασης γεωγραφικής ένδειξης. Ε, θέλουμε να ξέρουμε καλύτερα τι θα συνεπιφέρει. Και εγώ σε αυτή τη γραμμή λοιπόν θα κινηθώ. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής σας ε, προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνει ότι στόχος είναι να προστατευτούν τα αυθεντικά μη γεωργικά προϊόντα με βάση κάποιες παραγωγικές μεθόδους παραδοσιακές που, που τελούν πολιτιστική κληρονομιά μιας συγκεκριμένη γεωγραφικής περιοχής σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης καλωσορίζουμε και το ενδιαφέρον που δείχνεται για τη διατήρηση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και των σχετικών δεξιοτήτων. Επίσης, Με ικανοποιεί το γεγονό ότι θέλετε να ενημερώνετε καλύτερα καταναλωτέ για τη γνησιότητα των προϊόντων και για την προστασία των ε, νόμων ε, δικαιούχων και παραγωγών αυτών των καταχωρημένων προϊόντων. Σίγουρα υπάρχει και οικονομικό δυναμικό ε, στο σύστημα αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων για τη διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασία, για τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και για βελτίωση τη ελκυστικότητα διαφόρων περιοχών και ιδίω τουριστικών προορισμών. Εξού και θα ε, δώσουμε συνέχεια και θα δούμε αν μπορούμε να παρατείνουμε αυτό το σύστημα προστασίας ε, των γεωγραφικών ενδείξεων και αν το επεκτείνουμε και στα μη γεωργικά προϊόντα. Θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, ε, ιδίως ό,τι αφορά την ανάγκη να συνδυάσουμε την τεχνολογική καινοτομία με την ποιότητα και την γνησιότητα του τελικού προϊόντος. Είναι ανάγκη επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στη θέσπιση σαφών κανόνων όταν η ονομασία χρησιμοποιείται εκτός μιας συγκεκριμένης περιοχής, γιατί είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε και στην περιοχή αυτή προέλευσης, Και θέλουμε επίσης να λάβουμε υπόψη τις εφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις στα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε την αχρίαστη γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά την καταχώρηση αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων. Η πράσινη βίβλος έγινε θετικά αποδεκτή. Η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εξέφρασαν θετική άποψη θα λάβουμε υπόψη μα και τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ αυτών τη συστάσει τη ε, δική σα Επιτροπή για τι Γεωγραφικέ Ενδείξει και εν συνεχεία θα δούμε με ποιο τρόπο θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα είναι σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα η προσπάθεια την οποία έκανε ο συνάδελφος Διακόνου είναι μια πολύ καλή προσπάθεια τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνσης και θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοι ε, να ε, συζητηθούν. Πάντως, όπως είπε ο εισηγητής και σε συνεργασία με τους Κιώδης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσουμε ε, συνεργαζόμενοι θα επιστήσουμε και την προσοχή των κρατών μελών να αναγνωρίσουν την αξία κάποιων προϊόντων τα οποία συνδέονται με την τοπική γνώση και να τους πείσουμε για την αξιοποίηση αυτής της τεχνογνωσίας μέσω μιας καλύτερης αναγνώρισης και μέσω της χρήσης των ε, καινοτομιών. Όπως είπε ο συνάδελφος Διακόνου, το θέμα δεν είναι μόνο η παράδοση, αλλά και η καινοτομία. Λοιπόν, η έκθεση αυτή θα συζητηθεί στις 12 Μαΐου ε, στην Επιτροπή και τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Υπολογίζουμε λοιπόν στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Διακόνου. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα και σωστά. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι μελέτες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Να πω ότι στη δική μου περιφέρεια, στο δικό μου χωριό, όλα τα πύληνα τα έφτιαχνε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε την ικανότητα σε ένα συγκεκριμένο λόφο, από τον οποίο έπαιρνε τον πύλο του για να φτιάξει ακριβώς ε, τα προϊόντα του. Μετά από τη δεκαετία του 90 όταν υπήρξε μια κάποια ανεργία στην περιοχή, άρχισαν να κλείνουν τα εργοστάσια, ε, συζητούσα με κάποιους παλιούς μου συμμαθητές και μου λέγανε δεν ξέρω τι θα κάνουμε γιατί δεν έχουμε δυστυχώς δουλειές. Και τους ρώτησα, αυτός ο, ο άνθρωπος ο κεραμιστής είναι ζωντανός ναι, ναι, μου λένε ότι είναι μια χαρά και έχει 7 παιδιά και όλα τα παιδιά έφυγαν και πήγαν στις πόλεις. Δεν ασχολήθηκαν πια α, με... με τις κεραμικές αυτές θερμάστρες τις οποίες ε, ε, κατασκεύαζε στο παρελθόν. Τερακότα de cel mai înalt nivel, exact din dealul acela niciunul dintre oameni nu este copilul acelui bătrân care a murit. Και δυστυχώ κανένας δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δυνατότητα να φτιάχνει τους φούρνους αυτούς από κεραμικό υλικό. Δυστυχώ πέρασε. Η εποχή πέθανε ο, ο ιδιοκτήτης. Ίσως να έχετε δει ε, το έργο του Ταρκόφσκι Ρουμπλιόφ το πρόβλημα ήταν οι καμπάνες, ποιος ξέρει να φτιάχνει καμπάνες. Και είχε μείνει ένα παιδί μόνο το οποίο ήξερε να φτιάξει καμπάνες και γι' αυτό το παιδί η δραστηριότητά του ήταν χρυσορυχείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν θέλω να πω. Εγώ φοβάμαι ότι όλες αυτές οι γνώσεις θα χαθούν. Όλοι θα αγοράζουμε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ που δεν ξέρουμε ποιος τα έχει φτιάξει με λίγα λόγια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σεβαστούμε την Ευρώπη και τον πλούτο της, τον παραγωγικό, να τον διατηρήσουμε και να τον αναπτύξουμε. Di eh, mettere tutto questo nella, nella sua relazione e comunque la ringraziamo molto Σας ευχαριστώ λοιπόν και για το πάθος το οποίο επιδείξατε. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για τις νέες στρατηγικές για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι από το 2010 με τη συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός έγινε κοινοτική αρμοδιότητα και μέσω της αρχής της επικουρικότητας βέβαια. Ε, και έχουμε μία γνωμοδότηση σήμερα για την πρώτη έκθεση για τον τουρισμό της έκθεσης ε, της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Είχαμε και την πρώτη ανακοίνωση παλαιότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τουρισμό και νομίζω ότι ο πολιτιστικός ε, τουρισμός έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Ο συνάδελφος Μόργανο έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την ευτυχία που έχω να σα παρουσιάσω την έκθεση για τι νέε προκλήσει που μπορεί να αντιμετωπίσει ο τουρισμό στην Ευρώπη. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι πρέπει να περιοριστούμε στου 1500 χαρακτήρε για την σύνταξη του κειμένου και έτσι δεν είναι δυνατόν να είμαι εξαντλητικό. Θα κάνω όμω ό,τι μπορώ. Θα μπορέσετε βεβαίω να διαβάσετε ότι έχω, και θα διαπιστώσετε ότι έχω περιοριστεί μόνο σε νήξει για τα βασικά θέματα τα οποία θεωρώ πως μπορούν να αποτελέσουν μηνύματα κλειδιά για την Επιτροπή των Μεταφορών που είναι αρμόδια κατθήλην. Και περιορίζομαι στα εξή θέματα. Λοιπόν, καταρχάς την ε, κοινωνική, διανοητική και οικονομική σημασία του πολιτιστικού τουρισμού που αφορά άλλωστε την δική μας την ε, Επιτροπή ιδιαιτέρως, την ε, άκρο επίκαιρη πρόκληση του να εξασφαλίσουμε τρόπους εξασφάλιση του, της μεταξύ της επέκτασης του τουρισμού αλλά και της διαφύλαξη και αξιοποίηση και αναβάθμισης του πολιτιστικού μας ε, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ε, αλλά βέβαια και τη δημιουργία νέων, νέων ε, έργων τέχνης ή νέων τόπων επίσκεψης, γιατί μπορούμε πάντα βέβαια να προστατεύουμε και να προβάλλουμε το παρελθόν, αλλά πρέπει να κοιτάμε και προς το μέλλον. Επίσης θα πρέπει να προβάλλουμε, να δώσουμε κίνητρα για τον πολιτιστικό τουρισμό, όχι μόνο με βάση προγράμματα και πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με, πρόταση, με πρόθεση της ιδέας για νέα μέσα, που μπορούν να έχουν στα θέση τους οι πολίτες και ιδιαίτερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιστεύω και να υπογραμμίσουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό της ποιότητας Ποιοτικό τουρισμό λοιπόν με κεντρικό ρόλο την, ε, το ρόλο της ε, πολιτιστικής εκπαίδευσης. Γιατί ξέρουμε βέβαια ότι δεν είναι όλοι οι συμπολίτες μας εξοικειωμένοι με την αναγνώριση και εκτίμηση της κουλτούρας, του πολιτισμού, του πολιτιστικού έργου. Έτσι λοιπόν, Μπορούμε από πολύ νεαρή ηλικία, βέβαια στην, στο πλαίσιο τη οικογένεια, στον κόλπο, τη οικογένεια, αλλά και στο σχολείο, να δίνουμε κίνητρα και να ευαισθητοποιούμε. Γιατί χρειάζεται βέβαια και η σχετική εμπειρία πάντα για την, αξιοποίηση, για την αξιολόγηση και εκτίμηση του πολιτιστικού έργου. Ιδιαίτερα πρέπει να δοθούν ευκαιρίε σε όλου του πολίτε και πάνω απ' όλα σε εκείνου που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. οικογένειε με μικρά παιδιά, ε, άτομα με αναπηρίε, άτομα ηλικιωμένα για να μπορούν και αυτά με κάθε δυνατή διευκόλυνση να ε, μπορούν να χαίρονται τα πολιτιστικά αγαθά. Ένα παράδειγμα που θα σας δώσω είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε όχι μόνο τα αρχιτεκτονικά εμπόδια στην πρόσβαση στο πολιτιστικό αγαθό, αλλά και άλλου τύπου εμπόδια που μπορούν να δυσκολεύουν την πρόσβαση στο ε, πολιτιστικό αυτό αγαθό. Ιδιαίτερα λοιπόν προτείνω να γίνεται σωστή διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού, του ευρωπαϊκού πολιτιστικού αγαθού, ενός από τους κυρίους πλούτους της Ευρώπης και θέλω να πω ότι αυτή η πολιτιστική κληρονομιά είναι που καθιστά την Ευρώπη έναν από τους κύριους προορισμούς για τους ε, τουρίστες ε, σε όλο τον κόσμο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με 40% υπενθυμίζω στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι αν θέλουμε να διευκολύνουμε, να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία στα θέματα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και να διευκολύνουμε και να προσελκύσουμε περισσότερε ροέ τουριστών, πρέπει να βρούμε τη σωστή αυτή ισορροπία και να εντοπίσουμε στρατηγικέ που και θα προβάλλουν και θα διευρύνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό αγαθό και θα διαφυλάσει την πολιτιστική μα κληρονομιά. Με μερικά παραδείγματα θα ήθελα να καταστώ πιο σαφής. Υπάρχουν καταστάσεις αφόρητες αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά αφόρητες, που δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Φερειπίν τα τεράστια κλαζερόπλια στο λιμάνι της Βενετίας ή τα μιλούνια των επισκεπτών στο παλάτι της Αλάμπρα στη Γρανάδα ή τεράστιες εχμές προσέλευσης τουριστών στο Ντουμπρόβνικ ή αλλού ή στην Πράγα. Επίσης πρέπει να προβάλλουμε και να δώσουμε ε, κίνητρα για έναν πολιτιστικό τουρισμό προς τους ε, Ευρωπαίους πολίτες με έναν τρόπο που θα διευκολύνει την πρόσβαση. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει όπως έχουμε ακριβώς και την διεθνή ε, ταυτότητα των φοιτητών που έχει προαγάγει η UNESCO να έχουμε μια ευρωπαϊκή κάρτα πολιτισμού για τον Ευρωπαίο πολίτη με πρόσβαση και διευκολύνσεις ως προς την πρόσβαση στα μουσεία, τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς τόπους, τις βιβλιοθήκες, αρχεία και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο και μια πραγματική προστιθέμενη αξία για τον πολιτιστικό τουρισμό στην Ευρώπη. Για τους πολίτες μας πολύ σημαντική πρακτική υποστήριξη, αλλά ταυτόχρονα και ένα σημαντικό συμβολικό μήνυμα ότι όλοι είμαστε μέτοχοι της ίδιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και θέλω Κλείνοντα, μια και δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σημειώσω ότι μια και ήταν περιορισμένη η έκταση του κειμένου μου, θα καταθέσω εγώ τροπολογίε στο κείμενο ώστε να το εμπλουτίνω με τα θέματα που θα ήθελα. Θα κάνω αναφορέ σε υφιστάμενα ε, σχέδια που πρέπει να διατηρηθούν ε, και να ενισχυθούν ασφαλώς ε, θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες, οι πολιτιστικές διαδρομές της Ευρώπης, το πλαίσιο πολιτιστικής κληρονομιάς και το Creative Europe. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της ψήφιος που πρέπει να συνεχιστεί. Πρόκειται για πολύ σημαντική πτυχή. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ανήκει βέβαια στον κλάδο και της καινοτομίας και πρέπει να υποστηριχθεί γιατί υποστηρίζουμε με τον τρόπο αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θέλω επίσης να αναφερθώ και στην αναγκαιότητα να κάνουν μια προσπάθεια για να αναγνωριστούν οι λιγότερο γνωστές ίσως ζώνες πολιτιστικού ενδιαφέροντος που όμως πρέπει και αυτές να υποστηριχθούν. Σταματώ εδώ, περιμένοντας τις προτάσεις και τις συστάσεις των συναδέλφων. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να προσελκύσουμε, να διεκδικήσουμε τη μεγιστή δυνατή ε, προσοχή από τους συναδέλφους ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μόρκανο. Θα δώσω το λόγο στους ο κύριος πρώτο, πρώτος, στους Κιώδης. Ο κύριος Μοργκάνος συνέταξε ένα πολύ καλό κείμενο βάση που καλύπτει σε βάθος την πολιτιστική διάσταση του τουρισμού που κατά τη γνώμη μου αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης για την τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για τη δημιουργία των νέων τουριστικών προϊόντων, να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές θεματικές ε, διαδρομές ανά την Ευρώπη. Ο θρησκευτικό τουρισμό είναι μία από αυτέ. Η γαστρονομία, η εινολογία και ο αγροτουρισμό μία δεύτερη. Διάβασα πρόσφατα την ε, εξαιρετική έκθεση του κυρίου Φίσα. Η γαστρονομία αποτελεί κίνητρο για πολλού επισκέπτε και συνδέεται με τι παραδόσει μα. Και άλλο φυσικά η εκπαίδευση, τα θερινά προγράμματα και τα προγράμματα ανταλλαγή, κυρίω για τα παιδιά μα. Επιτρέψτε μου όμω να σταθώ ιδιαίτερα στι δυνατότητε του αθλητικού τουρισμού που μπορεί να αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους κλάδους τουριστικής ανάπτυξης και αφορά όλα σχεδόν τα αθλήματα. Κυρίως <clears throat> όσον αφορά τη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων και τη φιλοξενία συλλόγων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Ας μην ξεχνάμε πως ένα αθλητικό γεγονός αποτελεί πόλο έξι για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Τέλος, οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του τουρισμού, η καθοδήγηση των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων είναι καθοριστική και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αγαπητέ κύριε Μοργάνο, συγχαρητήρια και πάλι για το εξαιρετικό κείμενο που συντάξατε. Αντιλαμβάνουμε ότι οι περιορισμοί στην έκταση του κειμένου δεν βοηθούν στο να αποδώσουμε όπως θα θέλαμε όλες τις σκέψεις μας. Θα καταθέσω ορισμένες ε, τροπολογίες που θα κινηθούν στα πλαίσια που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. così. Eh, il collega Zambaschi? Zambaschi. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Η έκθεσή του παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, είναι δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο να παίξει στις τουριστικές δραστηριότητες, μπορεί να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 195 συγκεκριμένα της συνθήκης αυτά τα οποία μπορεί να κάνει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα κάνει σε εθελοντική βάση βέβαια. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και ε, με την τουριστική αυτή δραστηριότητα, τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε και εκτός Ευρώπης και η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι τεράστια και πρέπει πρώτον να τη διατηρήσουμε και μετά να την αναπτύξουμε. Πολλά είναι αυτά τα οποία έχουμε να επιδείξουμε και σε επίπεδο αρχαιολογικό και σε επίπεδο πολιτισμού γενικότερα και έτσι να προστατεύσουμε και την ποικιλότητα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οκτώ εκατομμύρια ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3,3% του ενεργού πληθυσμού και αν λάβουμε υπόψη μας και τους συνδεδεμένους τομείς όπως ε, τις οικοδομές, τις διανομές, τις μεταφορές κτλ. Ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει και τα 15 εκατομμύρια. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μιλάμε για θέσεις απασχόλησης. Η ανάπτυξη στον τομέα αυτό θα φέρει και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. η ποιότητα του τουρισμού είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιοχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι εκεί όπου δεν υπάρχουν καθορισμένα επίπεδα ποιότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πολλά να προσφέρει. Εμείς στην Βουλγαρία δεν έχουμε ας πούμε τέτοιου είδους ποιοτικά αναγνωρισμένα επίπεδα πέρα από το θέμα της βαθμολόγησης των ξενοδοχείων κτλ. Κάτι το οποίο πολλές φορές δεν γίνεται και με ικανοποιητικό τρόπο γιατί είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε, τον ψηφιακό κόσμο και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιουτσούκ έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μόργανο που τόνισε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια σχόλια. Η Ευρώπη πράγματι είναι ένας ε, πάρα πολύ σημαντικός πολιτιστικός τουριστικός προορισμός Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες ε, και από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες. Οι διεθνείς αφήξεις ε, αυξάνονται ε, βέβαια. Χάσαμε ένα μερίδιο της αγοράς γιατί αναδύονται νέοι προορισμοί από άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ποικιλία, την πολυμορφία του ευρωπαϊκού τουρισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, τεχνολογίες των πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε και την βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι επενδύοντας στον άνθρωπο ε, προωθούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα. Και πρέπει ε, να προσελκύσουμε περισσότερους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε το πολύγλωσσο κεφάλαιο, το εξειδικευμένο ανθρωπίνο κεφάλαιο. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε τη σημασία μακροχρόνιων επενδύσεων για την επίτευξη κάποιων τάσεων, σταθερών τάσεων, για την προστασία της ε, πολιτιστικής οικονομίας και βέβαια και του περιβάλλοντος. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων είναι επίσης σημαντικό. Η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, μουσείων, τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων επίσης πρέπει να προωθηθεί για να έχουμε καινοτόμα βιώσιμα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των τουριστών. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτιστική πολυμορφία. Αυτό πρέπει να τον λάβουν και οι διάφοροι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Γιατί πρέπει να προωθήσουμε τη μοναδικότητα, ε, την ιδιομορφία της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ. Ε, ε, η κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μόργανο για την έκθεσή του. Ένα σημείο θα σχολιάσω. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Το και ο κύριος ε, Κούτσικ ότι θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τα μεγάλα κρουαζερόπλια. Πηγαίνουν στα λιμάνια και εκπέμπουν ε, πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα σε περισσότερες ε, περιπτώσεις. Πραγματικά κατεπηγόντω πρέπει να προωθήσουμε τον εφοδιασμό των λιμένων ε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Και οι πολίτες το ζητούν. Αναστούν βιώσιμους τρόπους για τον πολιστικό τουρισμό. Για την Ελλάδα νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, το γνωρίζω. Τι μπορείτε να κάνετε για τα νησιά, αλλά και για άλλους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Και πραγματικά θα ήθελα να εστιάσετε σε αυτό το σημείο, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ευχαριστώ. Λέγα Σεντρόβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μόργαν για την ε, νομοδότησή του που προωθεί μια νέα προσέγγιση για τον τουρισμό και για τις μεταφορές. Μίλησε και για τον αθλητικό τουρισμό, πολύ σημαντικό. Για τον αθλητισμό μπορεί κανείς ε, να ταξιδέψει για να δει κάποια αθλητική διοργάνωση, αλλά και για να ασχοληθεί ο ίδιο με ένα άθλημα, και χάρη ποδηλατικοί αγώνε. Επίση, θέατρα και όλα αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και τις διόψεις του νομίσματος. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι παρέχουμε μια έκπτωση, δίνουμε μειωμένη τιμή, θα πρέπει να στοχεύουμε και στο σωστό κόσμο, ε, στους ε, ομάδες στόχους, νέες, ε, νέοι άνθρωποι, οικογένειες. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να, χαθεί, να χαθούν κάποια έσοδα, άρα θα πρέπει να αντισταθμιστεί αυτό. Πάντως πιστεύω ότι είναι καλό να προσφέρονται μειωμένες τιμές για κάποιες κατηγορίες κάποιες ομάδες πληθυσμού για να μπορούν να πάνε σε κάποιες διοργανώσεις, αλλά επαναλαμβάνω να καλύψουμε και την απώλεια εισοδήματος για κάποιες άλλες κατηγορίες πληθυσμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση του κυρίου Μοργκάνο ιδιαίτερα σχετικά με τις δυνατότητες του πολιτισμικού τουρισμού. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία όμως θα πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο, όπως η πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες. Όπως είπε ο κύριος Διακόνος, συνδέεται το θέμα του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ενθάρρυνση ε, των νέων τουριστικών δρόμων και δραστηριοτήτων. Έχουμε εδώ δυνατότητες για να προσελκύσουμε ε, κόσμο σε ε, περιοχές οι οποίες μπορεί να μην παρουσιάζουν τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον αλλά να δείξουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Σας ευχαριστώ και για αυτή την παρατήρηση, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Γι' αυτό θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μόργανο λέγοντας ένα πράγμα μόνο από πλευράς μου ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο αποτελεί αμετακίνητο ε, θα έλεγα ενεργό στοιχείο μιας περιοχής. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φύγει σε κάποια φάση. Μπορούμε λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε με καλό τρόπο. Το θέμα είναι πως θα μπορέσουμε να κερδίσουμε νέα κοινά, πως θα αυξήσουμε την περίοδο ενδιαφέροντος Νομίζω ότι αυτά είναι επιμέρους θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Να δούμε και τον ρόλο της ψηφιοποίησης, να δούμε επίσης τον τουρισμό σε σχέση με κάποια πολιτιστικά συμβάντα όπως οι εκθέσεις, οι μεγάλες, τα φεστιβάλ κινηματογράφου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ε, ε, μπορεί να βοηθήσουν, όπως και τα πολιτιστικά δίκτυα και οι πολιτιστικές διαδρομές είναι και αυτά αφορμές για αύξηση του τουρισμού και σε οικονομικό επίπεδο και να δούμε επίσης ε, και τα προβλήματα για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Έχουν υπάρξει κάποια πειράματα και στην Ιταλία, αποφασίστηκε την Κυριακή να είναι δωρεάν όλα τα μουσεία και αυτό οδήγησε στον τριπλασιασμό των εισόδων στα μουσεία τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ε, μια εμπειρία που μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και από άλλες χώρες. Να μην ε, υποτιμάμε ότι πολλοί κόσμος ε, αρνείται να πάει σε τέτοιου είδους ιδρύματα μόνο και μόνο για, για οικονομικούς λόγους. Επίσης τα τουριστικά επαγγέλματα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητά τους, να βελτιώσουμε τις ικανότητες τις οποίες έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Όλες οι παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν είναι παρατηρήσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη. Θα δοθεί περισσότερη προσοχή στο θέμα της αηφορίας, είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Ε, να δούμε όταν κάποιος ζητά την αύξηση των επισκεπτών, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην σπάσουμε την ισορροπία η οποία υπάρχει σε περιοχές αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια καλή βάση θα έλεγα έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Περιμένω λοιπόν και τις τροπολογίες σας. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρονική άνεση. 12 Μαΐου είναι η προθεσμία και η ψηφοφορία προβλέπεται στις 15 και 16 Ιουνίου αν θυμάμαι καλά. θα έχουμε την δυνατότητα λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις τροπολογίες οι οποίες έχουν, θα κατατεθούν. Λοιπόν, πράγματι να επιβεβαιώσω, λέει η Πρόεδρος, ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 15 Ιουνίου. Στην Επιτροπή ε, Μεταφορών θα ψηφίσουν το Σεπτέμβριο. Ε, λοιπόν, Έχουμε και κάποια άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Καταρχάς να πω ότι οι επόμενες συνεδριάσεις είναι 16 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 12 μέσα. Τώρα θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Τώρα μόλις ήρθανε μαθητές από σχολεία, προέρχονται και από την Ιταλία, συγγνώμη που δεν είμαι πολύ αντικειμενική εδώ. Πρόκειται για μαθητές με τους καθηγητές τους από το Ινστιτούτο του Μεοντεφέλτρο στο Σάσο Κολβάρο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να διαθώσουμε το σχολείο αυτό, το οποίο συγκεντρώνει μαθητές από μια ευρύτερη περιοχή και έχει γίνει τεράστια προσπάθεια και από τους διδάσκοντες. Τους ευχαριστώ για την επίσκεψη. Συγγνώμη αλλά τελειώνει εδώ η συνεδρίαση της Επιτροπής. Είχαμε μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι να πήρατε μια καλή ιδέα του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πέντε λεπτά εμείς θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών. Ε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κάμερεβερτ για να αναφερθεί για τον τριμερή διάλογο ε, για τα θέματα των τηλεπικοινωνιών. Intanto benvenuti e mi scuso con voi, speravo